Good, good morning. Good, good morning. Καλημέρα σε όλους. Παρακαλώ βρείτε μια θέση να καθίσετε. Έχουμε μεγάλες ε, λίστες ψηφοφορίας ε, και πολλά θέματα να ψηφίσουμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατό. Γι' αυτό παρακαλώ καθίστε. okay if anybody wants to... Ωραία λοιπόν, έχετε απόλυτη ελευθερία λόγου, αλλά εκτός της αίθουσας παρακαλώ. Ξεκινάμε τις ψηφοφορίες. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίζω ιδιαίτερα του εκπροσώπους της Επιτροπής Αλίας ε, σε αυτή την ε, κοινή ψηφοφορία. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Με μεγάλη χαρά συνεργαζόμαστε μαζί σας. Να δώσω το λόγο λοιπόν πρώτα απ' όλα στον κύριο Μάτο. Παρακαλώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή που μας ε, έχετε επιφυλάξει. Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Επιτροπής για τα Δικαίωμα των Γυναικών για αυτή την κοινή συνεδρίαση που ελπίζω δεν θα είναι η τελευταία. Από την πλευρά της Αλίας έχουμε κάποια στοιχεία που σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα που είναι η δραστηριότητα των γυναικών που εργάζονται στην Αλία. Είναι πολύ θετικό λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή την κοινή ε, συνεδρίαση και φυσικά έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας και πάρα πολύ δουλειά. Και φυσικά και τη μεγάλη αυτή ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω αν κάποιοι από τους ηγητές θέλουν να λάβουν το λόγο, κύριε Ρωμέρα. Ρωμέβα, όχι, δεν θέλετε το λόγο. Ας ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες λοιπόν. Ξεκινάμε με την τροπολογία 13, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται 16. Είναι κατά τμήματα ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, ε, αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 16. Πέρας ψηφοφορίας. Δεν λειτουργεί. Ξαναπροσπαθήστε. Ξεκινά ξανά η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 16. Έχουμε ένα επιπλέον άτομο από τους πρέσινους. Okay, wait a minute. Because they have all... Μισό λεπτό διότι είναι εντάξει είχαν υπολογίσει στο πρόγραμμα ότι πρέπει να υπάρχουν μόνο πέντε μέλη. αυτο είναι ο λόγος. Ωραία λοιπόν, για τρίτη φορά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα τη τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Αστειευόμασταν. Πάμε για τέταρτη φορά. Άρχεται η ψηφοφορία. And the Πέρας ψηφοφορίας. Όχι, δεν έχει τελειώσει η ψηφοφορία. Now is closed. Τώρα έχει τελειώσει. Εγκρίνεται. Και τώρα ξέρετε πώς να πατήσετε το κουμπάκι. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπερ προφορική τροπολογία Υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Ναι. Ε, έχω αντίρρηση για αυτή την προφορική τροπολογία. Ε, είναι το μέλλον ο κύριος και εγώ είμαι ο βοηθός. Υπάρχουν άλλα μέλη γιατί πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο μέλη και τώρα επειδή έχουμε κοινή επιτροπή πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα μέλη. Κάποιος άλλος που έχει αντίρρηση. Τότε λοιπόν θα ψηφίσουμε επί αυτής της προφορικής ε, τροπολογίας, τροπολογία 18 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε τη 18. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 18. And Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ καταπίπτει το δεύτερο τμήμα περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 26 την 25 συγγνώμη 26 λέει ο πρόεδρος ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 26 άρχεται ψηφοφορία The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ ε, προφορική τροπολογία υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία στην τροπολογία 32 όχι ψηφίζουμε 32 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται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 Πέρας ψηφοφορίας. Όχι ακόμα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα παρακαλώ να ξαναελέγξετε την 25 και την 26 ήταν να καλέσετε για ψηφοφορία για την 26 και μετά ζητήσετε έλεγχο για την 25 και δεν είμαι σίγουρος ότι έγινε ψηφοφορία για την 26. Λοιπόν, ξανακάνουμε την ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρος, για τις 25 και 26. Απλά για να είμαστε σίγουροι. Ελέγχουμε την 25. Άρχεται η ψηφοφορία για την 25. Πέρα ψηφοφορίας και ελέγχουμε για την 26. Άρχεται η ψηφοφορία για την 26. Πέρας ψηφοφορίας. 25 και 26. Λοιπόν, εγκρίνονται και οι δύο. Περνάμε στη τελική ψηφοφορία για το όλο ψήφισμα με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν στον συζητητέ. Ευχαριστούμε πολύ που βρίσκονταν εδώ. Hi. Um, Parvanova would like to make a short statement just before the vote, just for you to know.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 Okay, dear colleagues, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τώρα με τις ψηφοφορίες. Να ξεκινήσουμε με την έκθεση της κυρίας Παρβάνοβα για την βία κατά των γυναικών. Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια, τρία για τη λίστα ψηφοφοριών. Θα κάνουμε αυτή την ψηφοφορία λίγο πιο αργά, διότι τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα. Θέλω λοιπόν να έχετε το χρόνο να καταλάβετε πολύ καλά τι λέω. Αν πω κάτι περίεργο, παρακαλώ μην διστάσετε να με διακόψετε και να μου πείτε ότι έχω λάθος. Ήθελα να επισημάνω τρία πράγματα στη σελίδα 7. Λέει στη συμβιβαστική 18 λέει πηγαίνετε στην τροπολογία 114. Αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να πάτε στο ΛΥΜΠΕ 9. Με παρακολουθείτε? Το δεύτερο, στη σελίδα 14. Στο τέλος, Στη συμβιβαστική 6 λέει πηγαίνετε στην ε, τροπολογία 43. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να πάτε στην τροπολογία 45. 43 δεν είναι καν δίπλα. Η 45 ακολουθεί στην επόμενη σελίδα. Λέει go to, είναι μετά η τροπολογία αυτή. Λοιπόν, σελίδα 14, συμβαστική 6, επαναλαμβάνω, κομπ 6 και στη δεξιά στήλη βλέπετε εφόσον εγκριθεί μεταβείτε στην τροπολογία 43 αλλά ουσιαστικά είναι λάθος το 43 πρέπει να πάμε 45 και τέλος ε, μια τεχνική κατατμήματα ψηφοφορία για τη ΛΥΜΠΕ 5 στη τελευταία σελίδα και τα τμήματα έχουν χωριστεί σε λάθος σημείο. Εκεί που βλέπετε λέει calls on member states to properly ratify the convention. Εκεί γίνεται ο διαχωρισμός και το υπόλοιπο κείμενο είναι το δεύτερο κομμάτι. Τελευταία σελίδα στη λίστα ψηφοφοριών. Λίμπε 5. στο κείμενο κάτω κάτω στη σελίδα 25 στη σελίδα 25 κάτω κάτω στο κείμενο στη λίστα πιθανώς να μην το προσέξατε καν ε. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Παπανόβα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις ε, και όλους ε, όσοι εργάστηκαν σε αυτή την έκθεση. Ήταν μια δύσκολη πρόκληση. Είναι πρώτη φορά που η Επιτροπή μας ε, λειτουργεί με νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά με τη βοήθεια των συνεισηγητών και της γραμματείας καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το κείμενο και ελπίζω να είναι επιτυχής η έκθεση αυτή. Μια διευκρίνηση. Μην αποθαρρυνθείτε ε, από την σύνθετη λίστα ψηφοφοριών λόγω της διαδικασίας. Έχουμε πρώτα το ψήφισμα και μετά το παράρτημα. Διαφέρει από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Επίσης μην αποθαρρυνθείτε γιατί υπάρχουν πολλά μείον πολλαπλήν δεν σημαίνει ότι δεν ευθυγραμμίζονται με το σκεπτικό της έκθεσης, απλά ε, έχουν συμπεριληφθεί με άλλο τρόπο. Μην σας αποθαρρύνουν λοιπόν τα μείον, τα πλήν που θα δείτε, έχουν συμπεριληφθεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Απλά είναι ένας ε, περίεργος τρόπος αυτός της παρουσίασης της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Το συγγνώμη λοιπόν για οτιδήποτε αποθαρρυντικό μπορεί να αντιληφθείτε. Όλα έχουν συμπεριληφθεί, υπάρχει μια ισχυρή ε, ε, άποψη της Επιτροπής μας ε, με στιβαρές θέσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Ξεκινάμε την τροπολογία 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λίμπε 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε την 75 άρχεται η ψηφοφορία για την 75 πέρας ψηφοφορίας όχι ακόμα τρία μέλη λείπουν πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται Τροπολογία 76 με προφορική τροπολογία. Υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Όχι. ψηφισμού για την 76 λοιπόν. Ποιο είναι υπέρ. Ποιο είναι κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 126 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 78 υπέρ. Κατά αποχές λοιπόν, επαναλαμβάνουμε 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 80 καταπίπτει περνάμε στη συμβιβαστική 16 συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Ψήφι. Περνάμε στη ΛΥΜΠΕ 11, δεν έχει ψηφοφορία. Περνάμε τροπολογία 82, υπέρ, κατά, αποχές. Δεν ήταν σαφές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. The vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Λίμπε 15. Είναι κάποιο κατά τη προφορική τροπολογία. όχι. Να ψηφίσουμε για τη Λίμπε 15 υπέρ κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι 127 κατά πίπτη. Περνάμε στη Λίμπε 14 υπέρ κατά. Αποχέ. Να τσεκάρουμε τη Λίβε 14, ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is Πέρας φοφορίας It's rejected. Απορρίπτεται. Τροπολογία 84. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές να τσεκάρουμε την 88 άρχεται η ψηφοφορία της ψηφοφορίας σαφώς εγκρίνεται Τροπολογία 90 Κάποιο είναι κατά τη προφορική. Ε, όχι. Ψηφίζουμε για την 90 υπέρ. Κατά αποχέ. Απορρίπτεται. 89. Με προφορική, ε, είναι κάποιος κατά της προφορικής, όχι. Ψηφίζουμε την 89 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 93 δεν ψηφίζεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν 95, 96 και 92 καταπίπτουν. Περνάμε στην 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε έτσι στην 105, 105 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 δεν έχει ψηφοφορία συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ας περάσουμε λοιπόν στην 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Λίμπε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε. Να ελέγξουμε τα 130 ηλεκτρονικά αρχή ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 δεν έχει ψηφοφορία 135 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 135 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να περάσουμε λοιπόν ε, στην 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 2 υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίνεται αλλά για να είμαστε βέβαιοι ας τσεκάρουμε την 132 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 16 δεν έχει ψηφοφορία 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λίμπε 19 δεν έχει ψηφοφορία 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην επόμενη συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην επόμενη σελίδα συμβιβαστική 24 υπέρ κατά συμβιβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε στην τροπολογία 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία στην επόμενη σελίδα. Τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 καταπίπτει. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 10 στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 11 στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. συμβεστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε τροπολογία 70 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία στη συνέχεια στην τροπολογία 74 αντιρρήσει όχι ψηφίζουμε 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβεστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3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 118 ε, καταπίπτει 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 119 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε για όλο το ψήφισμα με ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας Εγκρίνεται καθαρά. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια στον... στην εισηγήτρια. Ωραία, προχωρούμε στην επόμενη ψηφοφορία. Σεξουαλική εκμετάλλευση και εκπόρνευση και αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων. Από τη συντάκτρια τη γνωμοδότηση είναι η κυρία Χάνιμπορ. Να σα επισημάνω ορισμένα σημεία του εγγράφου τη λίστας ψηφοφορία, μάλλον, γιατί είναι λίγο περίπλοκη και αυτή. Θα τα συζητήσουμε και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορία. Για παράδειγμα, υπάρχουν δύο τρόπολογίε με τον ίδιο αριθμό, κάποιες προφορικές τροπολογίες που λείπουν. Αλλά αυτά αφορούν σε περιπτώσεις που μάλλον θα, μα απασχολήσουν μόνο αν κάποιε συμβαστικέ τροπολογίες καταπέσουν, άρα πιθανότατα όχι. Δίνω λοιπόν τον λόγο στην κυρία Χάνιμπολ στην εισηγήτρια. Κυρία Χάνιμπολ, πρώτα πολύ σύντομα να πω ότι ήταν πολύ υποκοδομητική συζήτηση εχθέ και ευχαριστώ όλου και τους σκιώδει εισηγητές που βοήθησαν πολύ. Ευελπιστώ λοιπόν ότι θα το υπερψηφίσουμε το, στη γνωμοδότηση. Είναι σημαντικό το θέμα και ας μην χάσουμε την ευκαιρία να το ε, συζητήσουμε για να το ψηφίσουμε στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Σας ευχαριστώ όλους. Κυρία Κονελίσσα. Τρεις πολιτικές ομάδες έχουν ζητήσει αναβολή της ψηφοφορίας. Γιατί πράγματι είναι πολύ περίπλοκη ε, στα χάλια η κατάσταση ψηφοφορίας, λείπουν προφορικές τροπολογίες, υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες που αναφέρονται ως ταυτόσιμες ενώ δεν είναι, υπάρχουν προβλήματα στην αρρύθμιση, διπλές δύο φορές να, να καταγράφεται η ίδια τροπολογία. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίσουμε κατά πόσον χρειάζεται αναβολή της ψηφοφορίας. Από την πλευρά μας το ECR προτείνει αυτή την αναβολή. Η Γκούε επίσης, ο σκιώδης εισηγητής της Γκούε και οι σοσιαλιστές ζητούν να συνεχίσουμε, να, να ψηφίσουμε τώρα, σήμερα. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η θέση της Άλτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ προτείνω να ψηφίσουμε επί της αναβολής. Πρόεδρος, έχετε θεί λοιπόν θέμα διαδικασίας εάν θα ψηφίσουμε σήμερα ή όχι. Ε, θέλει κάποιο άλλο, η κυρία Γιανακουδάκη, κουκουδακη θελετε το λόγο επί τη ε, διαδικασία. Ναι, ναι. Είμαστε μία από τι πολιτικέ ομάδε που ανησυχεί γιατί εργαστήκαν αρκετά αργά το βράδυ το προσωπικό για να ετοιμάσει αυτή την κατάλογο ψηφοφορία. Αλλά όπω είπε και η Μέρη, εάν δεν ψηφίσουμε σήμερα, ε, είναι απίθανο να ψηφιστεί τελικά η γνωμοδότηση κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία. Μια και έχουμε ήδη εργαστεί, α ψηφίσουμε. Ε, υπάρχουν προβλήματα πράγματι, αλλά πρόκειται για γνωμοδότηση ιδίας πρωτοβουλία. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε να ψηφίσουμε, λοιπόν, πιστεύω. Κύριε Γκουμάη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκαθαρίσω κάτι για όλους. Έγινε μία συνάντηση των συντονιστών εχθές, δεν το έθεσε κανένας. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί αναφέρεται σήμερα, γιατί τίθεται σήμερα αυτό το θέμα. Θα έπρεπε να το είχαμε συζητήσει χθε στη συνάντηση των συντονιστών. Α μην υπονομεύσουμε το εξαιρετικό έργο τη ε, εισηγήτρια και όλων των συναδέλφων που προετοίμασαν αυτή την εξαιρετική αναφορά, την θέσουμε σε ψηφοφορία, γιατί διαφορετικά θα χαθεί. Και είναι εξαιρετικής ποιότητας, όπως και όλες οι άλλες. Κυρία Ζούμπερ. Η ομάδα της Γκουε θέλει να υποστηρίξει την πρόταση να ψηφιστεί τώρα η έκθεση αυτή, γιατί έχουμε κάνει όλη αυτή την εργασία. Χθε δεν έθεσε κανένα θέμα αναβολής είναι φανερό ότι είναι πολύπλοκος ο κατάλογος ψηφοφορίας, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε. Και στην προηγούμενη ψηφοφορία είχαμε προβλήματα, αλλά τα καταφέραμε. Η ομάδα μας έχει καθορίσει τη θέση της και τον κατάλογο ψηφοφορίας της. Επομένως, είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Παρβάνοβα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πολλές φορές στις συναντήσεις των συντονιστών είχαμε προβλήματα να αποφασίσουμε για τον τίτλο ή για άλλα θέματα που είχαν σχέση με τι γνωμοδοτήσεις, αλλά παλαταλίζαμε αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι καλύτερα να την αφήσουμε αυτή την ε, γνωμοδότηση για να μην υπονομεύσουμε την ίδια τη δουλειά μας. Ναι, και υπάρχει αυτή, αυτή αυτές τις διστάμενες απόψεις. απόψεις. Κυρία Χιμένες. Ε, Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ με αυτό που είπαν οι προλαλήσασες, οι συντονιστές. Νομίζω ότι είχαν κάνει μια συμφωνία, η συγγήτρια έκανε μια προσπάθεια συμβασμού σε ένα δύσκολο και πολύπλοκο θέμα. Βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος της θητείας. <clears throat> Ως εκ τούτου νομίζω θα ήταν πολύ σωστό να ψηφίσουμε. Και συμφωνώ με αυτά τα οποία ελέγχθηκαν για τα τεχνικά προβλήματα. Βέβαια δεν ευνοεί το έργο μας, αλλά δεν είναι σοβαρά αρκετά τα προβλήματα αυτά για να μας οδηγήσουν στην αναβολή της ψηφοφορίας. Εγώ θα προτιμούσα λοιπόν να ψηφίσουμε τώρα, ζυγίζοντας και τις δύο πλευρές, και είναι πιο σημαντικό αυτό από το να δώσουμε έμφαση στα τεχνικά προβλήματα. Κυρία Μορβάη. Πιστεύω ότι είναι ιστορική σημασία σε αυτή η γνωμοδότηση. Και υπάρχει μια δυναμική την οποία δεν θα πρέπει να τη χάσουμε. Γι' αυτό ας ψηφίσουμε τώρα. Κύριε Τελβό. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε τώρα την ψηφοφορία. Αλλά συμφωνώ και με την ε, σκιώδη ηγετρία του ΕΛΚ, η οποία προτείνει να την αναβάλουμε. Υπάρχουν ε, τεχνικά προβλήματα, μια και κάποιε τροπολογίε κατετέθησαν αργοπορημένα, που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ψηφοφορία την ίδια. Γι' αυτό και εγώ προτείνω να την αναβάλουμε. Πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει έχει τεθεί αυτή η πρόταση για αναβολή της ψηφοφορίας και πρέπει να την θέσω σε ψηφοφορία. Έχει δικαίωμα να αποφασίσει η Επιτροπή. Λοιπόν, ρωτώ, ποιοι είναι υπέρ τη αναβολής της ψηφοφορία. Κατά. Απορρίπτεται λοιπόν αυτή η πρόταση, άρα ψηφίζουμε σήμερα. Θα φροντίσω να προχωρώ αργά κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για να εξηγώ διάφορα θέματα ακόμα πιο αργά από ό,τι συνήθω. Ακόμα πιο αργά από ό,τι έκανα στην προηγούμενη ψηφοφορία. Λοιπόν, συμβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Που σημαίνει ότι πηγαίνουμε στην 66 και 67 οι οποίες είναι ίδιες. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτονται. 68. Ναι, βεβαίω, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικό έλεγχο 66-67, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. ψηφοφορία. Απορρίπτονται. Εξήντα Το υπέρ. Τροπολογία 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πηγαίνουμε τώρα στην συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά Ας την ελέγξουμε. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Στην 75 υπάρχει και προφορική τροπολογία. Υπάρχει ένσταση επί αυτή. Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε λίγο πρώτα για την 75. 75 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Α το ελέγξουμε αυτό. 77 άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. φορέ. Απορρίπτεται. Ναι, ε, ήθελα να επισημάνω ότι πάντα υπάρχουν τρία μέλη που δεν ψηφίζουν. Α, κατάλαβα, λέει ο πρόεδρος. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, λέει ο πρόεδρος στη γραμματεία. Ωραία, απορρίπτεται. 79. Δεν ψηφίζουμε επί της 78 γιατί έχει καταπέσει. Με εξαιτία τη συμβιβαστική 6. Το λέει τρεις γραμμές παραπάνω. Προχωρώ αργά, όπω βλέπετε. Στο σκιασμένο τμήμα της, ε, του καταλόγου ψηφοφορίας βλέπετε ότι η συμβιβαστική 6 προκαλεί, ε, ε, ε οδηγεί στο να καταπέσουν δύο τροπολογίε, 70 και 78. Άρα πάμε στην 79. 79 υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 80 υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. 70, 87. Η 86 καταπίπτει εξαιτία τη συμβιβαστική 8. Επομένω τώρα ψηφίζουμε για την 87. 87 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Να, να ελέγξουμε την ε, συμβαστική 10. Έναρξη της ηλεκτρονικής ψηφορίας συμβαστική 10. Πέρας ψηφορίας. Πρόεδρος, α, τώρα κατάλαβα. Υπάρχουν κάποια μέλη που, που, που δεν είναι παρόντα και έχουν αφήσει την κάρτα του. Εγώ νόμιζα ότι ήταν στο δωμάτιο και δεν μπορούσα να του ε, δω. Απλώ έχουν αφήσει το καρτελάκι του μέσα στο σύστημα ψηφορία. Αυτό ήταν όλο. Οκ. Okay. Ε, η 10. Τροπολογία 92. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Τροπολογία 92. Ηλεκτρονική ψηφοφορία έναρξη. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 93. Εδώ έχουμε τη ψηφορία κατά τμήματα. Για το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην 102. 102 τμηματική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε αυτό. Ε, έλεγχος λοιπόν για το πρώτο τμήμα της 102. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα πηγαίνουμε στην 109. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Ελεκτρονικό Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 113. 113 παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, κατά πίπτη λοιπόν 117, άρα 118. 118 υπέρ, κατά, εποχές. Ας την ελέγξουμε και αυτήν. Έναρξη ηλεκτρονικής φορές για την 118. Πέρας δεν Εγκρίνεται. 119. Τιματική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Για δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 120 ε, υπέρ. 1. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε αυτό. 121 λοιπόν. Ηλεκτρονική ψηφορία παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας φορείας Απορρίπτεται. Άρα 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 110, 123. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 124. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορία για την 124. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άρα πηγαίνουμε στην 127. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128 τμηματική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Υποχές. Εγκρίνεται για το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα της 128 έναρξη ψηφοφορίας. Σας ενημερώνω ότι ψηφίσαμε για την 127 ήδη. Τώρα είμαστε στην 128 στο δεύτερο της τμήμα. Γι' αυτό είναι. Σε αυτό αφορά η ηλεκτρονική ψηφορία που μόλις έκλεισε και εγκρίνεται. Τώρα, ζητώ συγγνώμη, κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλήσω κατά τη διάρκεια μια ηλεκτρονική ψηφοφορία, αλλά με ρώτησαν μια ερώτηση. 129 δεν τίθεται σε ψηφοφορία και πάμε στην 189. Υπέρ. Τα αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ Κατά. Από ποιες ελέγχουμε ηλεκτρονικά 130 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι, Α ελέγξουμε. 131, έλεγχος, έναρξη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 132, υπέρ. Κατά. Φοχέ. Ηλεκτρονικός έλεγχος, 132, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε στην συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 140, 140 υπέρ, κατά, εποχές. Κρίνεται 143 υπέρ, κατά, εποχές, Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 143. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρασε της Απορρίπτεται. Ε, επομένως ψηφίζουμε τώρα για την 144. 144. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίψετε. 145. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 146. Υπέρ. Κατά. Ε, εγκρίνεται. 147. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 153 τμήματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά η ηλεκτρονικός έλεγχος για την 155 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 156 υπέρ. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επομένως προχωράμε στην 161. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε, συγγνώμη, 168 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. αποχέ απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην 160, 176 μάλλον. Εδώ έχει κατατεθεί προφορική τροπολογία στην 176. Υπάρχει ένσταση όχι, άρα 176 μπορούμε να ψηφίσουμε. Α, ναι, συγγνώμη, δεν παρατήρησα ότι 176 έχει καταπέσει εξαιτία τη 18 τη συμβιβαστική, άρα 180. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 182. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 183. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 187. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 188 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα τρεις ίδιες τροπολογίες, Η 1, 2 και 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Δύο ίδιες τροπολογίες, Η 4 και η 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά ε, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 7, 11 και 14 είναι ίδιες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 ίδιες, η 9 και η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 17 έχει αποσυρθεί. 18 υπέρ. Κατά. εποχέ Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. εποχέ Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Α, ναι, να, να, βεβαίως να ελέγξουμε για την 19. 19 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε η ηλεκτρονική ψηφορία για την 21 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά εποχές Απορρίπτεται. 25 ε, κατά εγκρίνεται. 25 μάλλον έχει αποσυρθεί. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 και 33 είναι ίδιες. Υπέρ. Κατά. αποσχέσεις Εγκρίνονται. 32 υπέρ. Κατά. αποσχέσεις Εγκρίνεται. 34. 38. Και οι 55 είναι ταυτόσιμες και έχουμε τη πνευματική ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποσχέσεις. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 35. Τμηματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 τμηματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, 46 ε, την έχουμε ήδη καλύψει, την έχουμε ήδη ψηφίσει, επομένως τώρα ψηφίζουμε 47, 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50. Τμήματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Α, ωραία, ας ελέγξουμε για την 51. 51 ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ ψηφίστε. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56. Τμηματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Εγκρίθηκε. Τώρα. Συγχαρητήρια στην εισηγητή. Chair. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Κονέλ, σε έχετε το λόγο. Εν ώψη της ψηφοφορίας, ε, ορισμένα μέλη της Επιτροπής μας έχουν μια μειωνοτική μειονοτική θέση, η Ούριλη και Νούλετσεκ, Ρωμέβα Ιρουέδα, Κονέλσεν και Σοφίν Ινφέλτ των Φιλελευθέρων. Έχουμε καταθέσει μια άποψη μειοψηφία για την έκθεση αυτή. Θα καταγραφεί στα πρακτικά, λέει ο πρόεδρο, κυρία Νίμπλα. Σα ευχαριστώ κύριε πρόεδρε και εγώ έχω ακριβώ το ίδιο αίτημα. Εξ ονόματο τη κυρία Λούλινγκ, Κλά και εμού τη Ιδία θα καταθέσουμε μια ε, έκθεση μειοψηφία που θα έρθει σε εσά επί τη βάση του, της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του κανονισμού μας. Βεβαίως, λέει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόταση που θα μας δώσετε. Περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση. Αλλά θα δώσω τα το προεδρικό θόκον στην κυρία Στρέλα.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 Συνεχίζουμε με την έκθεση για την ισότητα ανδρών και γυναικών ή γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2012. 122 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε. Open the vote. Close the vote. Πέρας προφορίας. Απορρίφθηκε. Συγγνώμη, συγγνώμη, ήμουν αφηρημένη. Uh, amendment 126 and 27 and 28 are identical. In favour? Against? Abstention? Rejected. Απορρίπτονται. Ας ελέγξουμε αρχή την ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Rejected. Απορρίπτεται. Απο... 130 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε και πάλι άρχεται ψηφοφορία The Πέρας. Απορρίπτονται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Uh, The vote is closed. Πέρασε φοφορίες. Απορρίπτεται. 131. Υπέρ κατά εγκρίνεται 133 <clears throat> υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται εκπίπτει η 134 135 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστή 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε για την 139. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 143. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 147. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 149. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 και 163 που είναι ταυτόσιμες ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος για την 165. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται, 181 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται, 183 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται, 184 υπέρ κατά αποχές έλεγχος είναι 184 Άρχεται η ψηφοφορία. <clears throat> Πέρας. Εγκρίνεται. 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, θα σε ελέγξουμε όμως. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα Εγκρίθηκε. 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 190 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 191 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 202. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 205. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 207. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 208 υπέρ κατά συγγνώμη και πάλι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 210 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα εκπίπτει 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 216 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2-23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.30 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα εκπιτη 2.31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.34 <coughs> υπέρ κατά χέρι εγκρίνεται 2.67 υπέρ κατά χέρι συγκρίνεται συμβαστική 21 υπέρ κατά χέρι συγκρίνεται συμβαστική 26 υπέρ κατά χέρι εγκρίνεται Τροπολογία 235 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.37 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω άρχεται η ψηφοφορία επαλήθευσης Τη 237 ψηφίσουμε, Μαρία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Εκπίπτει 238 και η 39 επίσης. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 243. Ψήφι υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.59. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 2.65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Γιατί 265 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 266 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για 266 άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτει. 268 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 272 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 271 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2,70 εκπίπτει. 2,69 εκπίπτει. ...2,75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 276 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.88 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.93 υπέρ όχι δεν εκπίπτει, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 2, 94 και 95 εκπίπτουν, Συμβαστική τροπολογία 24. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 306. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 307 υπέρ. 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε. Άρχεται την ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 308 υπέρ κατά αποχές δεκτή 310 υπέρ κατά αποχές δεκτή 311 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 314 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 315 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ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 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είκοσι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 31 υπέρ κατά απόχειας εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά απόχειας εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά απόχειας εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά απόχειας εγκρίνεται. Σύμβαση 3 34 έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία επαλήθευσης. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57. Μια στιγμή. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνε απορρίπτεται συγγνώμη 64 ναι κυρία Παρβάνοβα μα δεν αναφέρεται ότι οι 53, 54 και 55 εκπίπτουν λόγω της συμβαστικής 5 και ούτε καν τις ψηφίσαμε. Ναι, πήγαμε στην τροπολογία 57 κατευθείαν. Έχετε δίκιο, μεγάλο το δίκιο σας. Θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες 53, 54 και 55 που ταυτίζονται. Μάλιστα. υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκαν έλεγχος, έλεγχος, εντάξει, άμα θέλετε άρχεται η ψηφοφορία έλεγχου πέρας απορρίπτονται πράγματι Πού ήμασταν τώρα. Ψηφίσαμε την 65. Ψήφισα υπέρ, λέει κυρία Μπάστου. Εγκρίνεται τότε, εγκρίνονται τι τροπολογίε αυτέ οι επίμαχε. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 65. Όχι, όχι, 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73. Κυρία Ντελβό. Δεν ε, ακούγεται κυρία Ντελβό. Έλαβε το λόγο με δίχως μικρόφωνο. Απερίφθη 67 ή όχι. ζητά έλεγχο η κυρία Ντελβό. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 67. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται. 73. Τροπολογία 73. Υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται 77. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 78. Υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 86 πέρας Απορρίπτεται. Συμβαστική 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 110 σε δύο τμήματα το πρώτο τμήμα έχει εκπέσει, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία τώρα, ηλεκτρονικά την ψηφοφορία. The Πέρας. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στην κυρία Ζουμπέρ. the oral question. Uh, on behalf of the committee. για την εξάλληψη των κριτηρίων των γενικών οργάνων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 Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 13 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή τον κύριο Γκούσταυσον, τον πρόεδρό μας. On behalf, yes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 Συνεχίζουμε με την τελευταία ψηφοφορία, την εξέλιξη των βασανιστήριων στον κόσμο. Να ρωτήσω από την κυρία Γιαναπουδάκη αν θέλει να πάρει το λόγο, συγγήτρια. Εκτός μικροφώνου, η κυρία συγγήτρια. Ενδιαφέρον ε, το σχόλιο της συγγήτριας, λέει ο πρόεδρος. Ξεκινάμε με την τροπολογία 9 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 9. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Να ελέγξουμε και το δεύτερο τμήμα, ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Καταπίπτει. Περνάμε στη συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρινέται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρινέται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρινέται. 17. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 22. Προφορική τροπολογία υπάρχει. Υπάρχει αντίρρηση. Όχι. Ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 επίσης, με προφορική τροπολογία υπάρχει αντίρρηση. Όχι, ψηφίζουμε 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 25 επίσης, έχει προφορική τροπολογία, υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 σε δύο τμήματα το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε την 31 το δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας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 Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται καθαρά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. So, and then we have the last... Έχουμε το σημείο 13 για την Κροατία και την Ουγγαρία. Δεν θα το συζητήσουμε θα αποτελέσει κομμάτι η έκθεση αυτή της διαδικασίας. Και περνάμε στο τελευταίο σημείο. Το 20 και τα διάφορα κάποια ενημέρωση για το νέο ε, χρονοδιαγράμμα για τις συναντήσεις μας το 2014 και το τελευταίο σημείο 21, επόμενη συνάντηση 12 Φεβρουαρίου 2014 από 9 μέχρι 12.30 και από 3 μέχρι 6.30. Εδώ ολοκληρώνεται η συνάντηση αυτή.